διορθώσεις εάν εντός 24 ώρου δεν διαφωνήσει μια πολιτική ομάδα τουλάχιστον 40 βουλευτές. Τα κείμενα θα τα βρείτε στο Seance on Direct και τις επικεφαλίδες τους θα δημοσιευθούν στο συνοπτικά πρακτικά. Ο κύριος Αλεξάνδρ Μίσκι ζήτησε ε, υπεράσπιση της ε, κοινοβουλευτικής του ασυλίας. Σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 του κανονισμού διαβιβάζεται